<coughs> Bien, euh, και κύριοι, συνάδελφοι, να αρχίσουμε την σημερινή μας συνεδρίαση, η οποία περιλαμβάνει λιγότερα θέματα από ό,τι είχαμε αρχικά προβλέψει. Βασικά δεν θα συζητηθεί το θέμα που αφορά την Ουκρανία, όπως είχαμε προβλέψει, διότι οι συνομιλητές μας είχαν κάποιο πρόβλημα. Άρα Έχουμε δύο θέματα στην ημερησία διάταξη. Το πρώτο αφορά το κέρες τη Αφρικής και ιδιαίτερο στην ε, αποστολή UCAP Nestor και ενημέρωση για την αποστολή της Υποεπιτροπής μας της προηγούμενης εβδομάδας και μετά θα συζητήσουμε την ε, ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία μηνάς που θα ζητήσουμε με τον κύριο Τοκάσκι. Έχουμε μαζί μας την τιμή να έχουμε τον στρατικό ε, Ζανβιέ, ο οποίος είναι διευθυντής της CPCC και τον κύριο Ετιέν Ντοπονσής, η κεφαλής της αποστολής. Η αποστολή ιου Νέστορ είναι η τελευταία από τις αποστολές στα πλαίσια της πολιτικής ε, εξωτερικής ε, και συνεργασίας του CDCC. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πρώτα απ' όλα την πιο σημαντική στην περιοχή αυτή, την, ε, επιστολή, ε, την αποστολή Αταλάντη. Έχουμε επίσης την αποστολή κατάρτισης της Σομαλίας που άρχισε από την Ουγγάντα και είναι τώρα στο Μογκαντήσιο με Ιταλό διοικητή, πρόκειται για στρατιωτική αποστολή και μία μη στρατιωτική αποστολή, την ε, UCAP Nestor, που τέθηκε σε κίνηση το 2012, πρόκειται, επαναλαμβάνω, για μη στρατιωτική αποστολή για την ε, ανάπτυξη των περιφερειακών ε, ναυτικών δυνατοτήτων και υποδομών στην περιοχή. Πρόκειται για μια ευρύτατη αποστολή. Δεν είναι πάντα προφανές το ότι θα μπορέσει να ε, βρει την ε, κανονική της πορεία στα πλαίσια όλων των ε, αποστολών που αναπτύσσονται στην περιοχή. Πρέπει να βρει τον χώρο στον οποίο θα αναπτυχθεί, χώρο που θα της αφήσει η Αταλάντη να πληρώσει. Ε, ο κύριος Λίζε και ο κύριος Σοφοκλέου, ο κύριος Τάραντ και εγώ πήγαμε στο Τζιμπουτί στα πλαίσια των ε, επαφών που θέλαμε να κάνουμε με τις αρχές του Τζιμπουτί πριν από μία εβδομάδα. Πάρα πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν, πάρα πολλά, τόσα πολλά που πραγματικά νομίζω ότι μπορούν ε, να αναπτύξουν δραστηριότητες πάρα πολλοί φορείς. Σήμερα λοιπόν εσείς, επικεφαλής της αποστολής, θα μας πείτε ποια είναι η δική σας άποψη, το δικό σας πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπετε τις αστέρτες του αναπνίξει αυτή η αποστολή. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ξέρετε πόσο επικριτικός πολλές φορές είμαι σε αυτές τις μη ε, στρατιωτικές αποστολές, αλλά κάτι το πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, το οποίο είδαμε στην αποστολή μας είναι η δυνατότητα που έχει αυτή η αποστολή να ε, παράσει εξοπλισμό. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο προξένει στον ενδιαφέρον ότι σε πολλά μέρη στα οποία πάμε και έχουν αναπτυχθεί τέτοιου είδους μη στρατιωτικές αποστολές, αυτό το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο πρόβλημα και για τους δικαιούχους είναι ότι μετά από την κατάρτιση που γίνεται δεν παρέχεται και ο απαραίτητο εξοπλισμό. Πράγμα που διαπιστώσαμε ιδιαίτερα στην Ήγυρα. Αυτή τη φορά λοιπόν είδαμε ότι υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα και θα δούμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί και σε ποιες ανάγκες μπορεί να ανταποκρίνεται. Πρόκειται για μια αποστολή λοιπόν η οποία αναμφίβολα εξελίσσεται σταδιακά και με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να μας πείτε εσείς κατά την άποψή σας, ποια είναι η αντίληψη των τοπικών φορέων και αρχών που ενδιαφέρονται αλλά πολλές φορές δύσκολα μπορούν να συγκεκριμενοποιήσουν τις ανάγκες τους και είναι και αντιμέτωποι με όλους αυτούς τους διάφορους φορείς τους εμπλεκόμενους. Κατά την άποψή σας πρόκειται για μια αποσκοτολή η οποία είναι αναγνωρίσιμη και μπορεί να είναι για όλες τις χώρες αυτές τις οποίες θα αναπτυχθεί χρήσιμη. Όλα αυτά τα θέματα θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε μετά από την παρουσίασή σας. Πώς θα προχωρήσουμε. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Ζερά ε, Ζανβιέ και μετά ο κύριος Ετσιέν Ντεποσέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε στην Αφρική δύο ε, στρατηγικές πολιτικές. Η δεύτερη είναι αυτή η UCAP Nestor στα πλαίσια Τη πολιτική που θέλουμε να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε την πειρατεία ιδιαίτερα και ιδιαίτερα στην περιοχή των χωρών κέρατο της Αφρικής. Πρόκειται για μια αποστολή που συμπληρώνει την Αταλάντη και την ε, ε, στρατιωτική αποστολή στην Σομαλία, καθώς και τα άλλα προγράμματα, τις άλλες πρωτοβουλίες, ε, τις οποίες έχουν αναλάβει ευρωπαϊκοί φορείς ή φορείς άλλες στα πλαίσια διεθνών οργανώσεων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μιλών, η Γιούκα Καπνέστορ μπόρεσε να παγιώσει την παρουσία της και να αυξήσει σημαντικά τις δραστηριότητές της στους πλέον σημαντικούς πυλώνες της ζώνης, στα πλαίσια της επιχειρησιακής της ευθύνης. Τα προσωπικό ε, που δραστηριοποιείται εκεί αυξήθηκε, το περιφερειακό γραφείο άνοιξε στην Σομαλιλάντ και ένας αξιωματικός συνδέσμου υπάρχει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στην Ταζανία. Στα πλαίσια της αποστολής λοιπόν αυτής στις 18 Μαρτίου επιβεβαίωσαν την στρατηγική που θα ακολουθηθεί. Έγινε εκτίμηση της στρατηγικής την οποία θα ακολουθήσει, των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει και η Γιούκα Νέστορ είπαμε ότι μπορεί στο μέλλον, στο άμεσο και στο μεσοπρόθεσμο, να μας επιτρέψει να εγγυηθούμε την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταπολεμήσουμε την πειρατεία στην περιοχή. Τα κράτη-μέλη πρέπει να πω ότι συνέστησαν ιδιαίτερος να επανεστιάσουμε την δέσμευση της UCAP Nestor στην Σομαλία υποστηρίζοντας όλους ιδιαιτέρως ε, τις δυνάμεις ασφαλείας στις παράκτιες περιοχές σε μια πολιτική διαφορετικών φάσεων, ώστε όταν ε, πληρούνται τα διάφορα κριτήρια σε θέματα ασφαλείας να υποστηρίξουν στην θαλάσσιο ε, περιβάλλον όλους τους κανόνες ασφαλείας και να υποστηρίξουν την ακτοφυλακή. Η στρατηγική αναθεώρηση επίση πρέπει να πω ότι συνέστησε την συνέχιση των δραστηριοτήτων τη αποστολή στι Σεϊχέλε και στο Τζιμπουτί και μια προοδευτική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στην Τανζανία. Δεδομένου ότι οι αρχές της Κένιας προς το παρόν δεν έχουν παράσχει την απαραίτητη πολιτική υποστήριξη, αποφασίστηκε οι δραστηριότητες στην Κένια να μην αναπτυχθούν περαιτέρω δεδομένου ότι δεν υπάρχει σαφή δέσμευση εκ μέρου κυβέρνηση αυτή. Αντιθέτω, τα κράτη-μέλη ζήτησαν η αποστολή αυτή να μπορέσει να αντιδράσει τάχιστα για να μπορέσει να θέσει σε εφαρμογή δραστηριότητε τα εάν οι αρχές της Κένιας επανέλθουν στην ε, πολιτική τους σε θέση το θέμα αυτό. Αποφασίστηκε εξάλλου να αναπτυχθεί και να υπάρξει στην ε, αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιεμένη ένας αξιωματικός σύνδεσμος Δεδομένου ότι η Εμένη ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το θέμα αυτό της καταπολέμησης της ε, πειρατείας και ε, συμμετέχει σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται για να την καταστολή της πειρατείας. Η αποστολή αυτή βρίσκεται σε βάση αναθεώρησης ε, των, στρατηγικών της σχεδίωσης ώστε να μπορέσει σύμφωνα με τις διάφορες ε, ενδείξει που γυλάβει από τα κράτη-μέλη να προσαρμόσει τη στρατηγική που θα κορίσει προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία του κατάλληλου βήματο όσον αφορά την ασφάλεια και την διοικητική υποστήριξη ώστε να υπάρχει μόνιμη ανάπτυξή της και παρουσία της στο Μογκαδίσιο της Σομαλίας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω και να σας παρουσιάσω την UCAP Nestor, την αποστολή αυτή, η οποία αναφίβολα είναι λιγότερο γνωστή από τις δύο άλλες στρατιωτικές αποστολές, οι οποίες δρούν στο κέρας της Αφρικής. Όμως, όπως θα σας δείξω, η UCAP Nestor συνεργάζεται άμεσα και πλήρως με τις άλλες δύο αποστολές. Πρόκειται για μια αποστολή πρόσφατη, μια που άρχισε τον Ιούλιο του 2012. Το 2014 λήγει η πρώτη εντολή που όπως είπε και ο στρατηγός Ζαβιέ θα παραταθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2016 κατά πάσα πιθανότητα. Η αποστολή λοιπόν του Nestor γράφεται στη γενικότερη προσέγγιση που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το κέρας της Αφρικής. Είναι μια ιδιαίτερη βέβαια περιοχή μια περιοχή για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέλησε να εντοπίσει συγκεκριμένα εργαλεία δράσης. Από την άλλη, δουλεύουμε στα πλαίσια της κοινή πολιτικής υπό την ύπατη εκπρόσωπο, αλλά και υπό τον πρέσβη Ρόντο, που είναι ο ειδικό μας απεσταλμένος στο κέρας της Αφρικής. Και είμαστε βέβαια πάντα υπό τον πολιτικό έλεγχο των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ναϊρόμπι πρώτα απ' όλα και στη Σομαλία. Συνεργαζόμαστε επίσης και είμαστε σε συντονισμό με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι υπάρχει συνοχή ανάμεσα στα διάφορα μέσα που χρησιμοποιούμε. Η αποστολή λοιπόν UCAP Nestor γεωγραφικά είναι μεταξύ της Αταλάντης και της UTM. Δηλαδή η Αταλάντη είναι στη θάλασσα εξορισμού και πέτυχε πολύ σημαντικά αποτελέσματα για την καταπολέμηση της πειρατείας, μια που πολλά σκάφη που ήταν θύματα πειρατείας ε, νιώθηκαν στον αριθμό. Η αποστολή λοιπόν Αταλάντη ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτή την άποψη. Από την άλλη μεριά λοιπόν υπάρχει η EUTM που είναι η στρατιωτική αποστολή της Σομαλίας και εμείς που είμαστε εμεί στρατιωτική αποστολή, είμαστε στη μέση και σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τον έλεγχο στη θάλασσα και στις ακτές. Και αυτό για πέντε χώρες που είναι στην περιοχή για το Τζιμπουτί, τη Σομαλία βέβαια, Τανζανία, Κένια και Σεχέλες. Γεωγραφικά λοιπόν αυτό είναι το πεδίο δράσης μας. Οι ακτές και τα ύδατα αυτών των χωρών του κέρατος της ε, Αφρικής. Πολιτικός μας στόχος είναι να επιτρέψουμε στις πέντε αυτές χώρες να ελέγχουν οι ίδιες τον θαλάσσιο χώρο τους και τις ακτές τους. Και έτσι μπορούμε να δώσουμε μια τελική λύση στο πρόβλημα της πειρατείας. Γιατί αν μπόρεσε να μειωθεί η πειρατεία στη θάλασσα, χάρη στις συνδυασμένες προσπάθειες των δυνάμεών μας, οι πειρατές παραμένουν όμως στην, ε, στο έδαφος και η Σομαλία είναι μια χώρα που εδώ και 20 χρόνια δρούν οι πειρατές και οι γείτονες χώρες δεν καταφέρνουν να ελέγξουν το θαλάσσιο χώρο τους αν υποθέσουμε ότι ελέγχουν την επικρατειά τους, την υπόλοιπη. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που έχει τέτοια περιφερειακή αποστολή η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δημιούργησε στην αρχή διάφορες δυσκολίε για το πώς θα λειτουργήσει η αποστολή, η αποστολή αυτή, γιατί είναι περιφερειακή, δηλαδή δράσει σε διάφορες χώρες, χώρες μάλιστα που είναι διαφορετικές μεταξύ του. Η Σεχέλης, για παράδειγμα, είναι μια ανεπτυγμένη χώρα, ενώ η Σομαλία από την άλλη είναι μια χώρα μοιρασμένη. Η αποστολή μας λοιπόν σήμερα έχει κάπου 100 εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 17 ευρωπαϊκές χώρες. Συμμετέχει και η Νορβηγία. Μάλιστα πριν από λίγες εβδομάδες προσλάβαμε και ντόπιο προσωπικό στο Τζιμπουτί ιδιαίτερα αλλά και στην Κένια. Σήμερα έχουμε λοιπόν 54 μέλη στο Τζιμπουτί, 16 στην Κένια, 6 στις Εχέλες και ένα άτομο στην Τανζανία. Η δομή της αποστολής έχει ως εξή. Υπάρχει το στρατηγείο το οποίο βρίσκεται στο Τζιμπουτί και μάλιστα είχαμε την τιμή να το επισκεφθούμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και από το Τζιμπουτί ελέγχουμε το σύνολο της αποστολής. Στην Κένια έχουμε ένα γραφείο όπου δεν εδρεύει η ομάδα που ασχολείται με την Κένια, γιατί δυστυχώς στην Κένια δεν μπορέσαμε να αναπτύξουμε δραστηριότητες, αλλά παρακολουθεί τα θέματα της Σομαλίας από το Ναϊρόμπι. Το Ναϊρόμπι είναι ουσιαστικά η είσοδο για τις δραστηριότητες στη Σομαλία. Και αυτό γιατί από το Ναϊρόμπι είναι που μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πτήσεις, easy flights, με την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Ναϊρόμπι και από εκεί μπορούμε καλύτερα να ελέγχουμε την κατάσταση στην Σομαλία. Στις Σεχέλες έχουμε μια, έχουμε μια έδρα που ασχολείται με τα θέματα της Σεχέλες και στην Τανζανία επίσης. Ο προπολογισμό είναι 23 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 2 εκατομμύρια περίπου για τον εξοπλισμό. Και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Το χρονοδιάγραμμα είναι ότι αρχίσαμε τον Ιούλιο του 2012 την αποστολή αυτή και ένα πρώτο στάδιο λύγει τον Ιούλιο και θα αρχίσει νέα εντολή από τον Ιούλιο του 2014 μέχρι κατά πάσα πιθανότητα το Δεκέμβριο του 2016 για να ευθυγραμμιστεί η αποστολή UCAP Nestor με εκείνη της Αταλάντης. Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητές μας τώρα. Να ενισχύσουμε την ικανότητα των χωρών αυτών να αντιμετωπίσουν την πειρατεία. Κύριος στόχος μας είναι να ενισχύσουμε το κράτος δικαίου και τις ικανότητες των χωρών αυτών από τη στιγμή που εντοπίζεται ένα δίκημα μέχρι την δίκη σε δικαστήριο. Προσπαθούμε δηλαδή να καλύψουμε όλο αυτό το φάσμα από το αδίκημα μέχρι τη δικαιοσύνη. Οι περισσότεροι πειρατές συνήθως τα αποδεικτικά τα πετάνε στη θάλασσα. Όταν λοιπόν δικάζονται οι πειρατές είναι δύσκολο να έχουμε αποδεικτικά στοιχεία. Προσπαθούμε λοιπόν να βοηθήσουμε σε αυτό με την ακτοφυλακή η οποία συλλέγει τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία από τη θάλασσα. Ο στόχος μας είναι βέβαια να προσαρμοζόμαστε κάθε φορά και στις ανάγκες. Οπότε ακούμε τι ζητούν οι χώρες και προσαρμόζουμε το πρόγραμμά μας ανάλογα με τη χώρα που καλύπτουμε. Η μέθοδός μας είναι η μέθοδος της συμβουλευτικής, δηλαδή δεν είμαστε εκτελεστικό όργανο, συμβουλεύουμε, εκπαιδεύουμε, καταρτίζουμε Βοηθούμε δηλαδή στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτών που εκπαιδεύουμε. Έπειτα παθεί και το νομικό πλαίσιο, γιατί υπάρχει και το νομικό πλαίσιο, ο νομικός πυλώνας, ο οποίος καλύπτει τους εισαγγελείς, τους δικαστές, αλλά και γενικά την δικαιοσύνη. Την νομοθεσία, για παράδειγμα, που εφαρμόζεται προκειμένου να καλύπτει αυτή και τα δικήματα της πειρατείας και να είναι αποτελεσματική στα αποτελέσματά της. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε πριν και είναι πολύ σημαντικό στον εξοπλισμό. Μπορούμε να προσφέρουμε εξοπλισμό. Βέβαια είναι μεγάλο θέμα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να την έχουμε αυτή τη δυνατότητα γιατί το ζητούν και οι χώρες που υποφελούνται. διότι αν η αποστολή μας δεν έχει έναν ελάχιστο εξοπλισμό, τότε τίθεται θέμα αξιοπιστίας μας. Έπειτα είναι και λογικό αν έχουμε μια ακτοφυλακή και θέλουμε να παρεύει σε ένα σκάφος και αν τελικά η ομάδα αυτή του Τσιμπουτή της Εχέλες δεν έχει τον εξοπλισμό που χρειάζεται για την επικοινωνία, για σωσίβια, τότε καταλαβαίνετε ότι η αποστολή ε, μειώνεται σε αποτελεσματικότητα. Άρα λοιπόν χρειάζεται εξοπλισμός. Είπαμε έχουμε ένα με δύο εκατομμύρια ετησίως για τον εξοπλισμό μας είναι λίγο, αλλά θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θέλουμε να το διατηρήσουμε αυτό. Είτε πρόκειται για κιάλια που βλέπει κανείς τη νύχτα, είτε πρόκειται για λεξίσφαιρα γυλαίκα, μέσα επικοινωνίας κτλ. Όλα αυτά πρέπει να ξέρετε ότι οι συνομιλητές μας στις χώρες αυτές τα εκτιμούν όλος ιδιαίτερος. Τώρα γεωγραφικά, για να περάσω περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούμε να διακρίνουμε τις χώρες όπου είχαμε ήδη σημαντικά αποτελέσματα μέχρι σήμερα και τις άλλες όπου είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και θα αναφερθώ όλος ιδιαίτερο στη Σοβαλία. Ε, και Τζιμπουτή πρώτα απ' όλα είναι οι χώρες στις οποίες έχουμε προχωρήσει περισσότερο. Η γενική στρατηγική της αποστολής ήταν να παρεμβαίνουμε πρώτον εκεί που είναι πιο εύκολο, γιατί για να έχουμε αποτελέσματα, για να έχουμε αποδείξεις, επιτυχίας που να μπορούμε να παρουσιάσουμε στις άλλες χώρες της περιοχής και σιγά σιγά προσπαθούμε να προσεγγίσουμε στην καρδιά του προβλήματος της πειρατείας που είναι βέβαια η Σομαλία και μέσα στη Σομαλία πιο συγκεκριμένα στο Πούκλαντ και το Καλαντό. Στο Τζιμπουτί λοιπόν μας ζητάνε την UCAP Nestor. Είμαστε εκεί εδώ και πάνω από δύο χρόνια. Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Είχαμε διάφορες δράσεις, έχουμε πυρογνώμονες που συμμετέχουν στην ακτοφυλακή ή στο ναυτικό των χωρών του Τζιμπουτί και των Σεχελών που συνομιλούν με τους ομολόγους της εκεί. Έχουμε για έναν ειδικό στο Υπουργείο, στο Τζιμπουτή, δικαιοσύνη για την νομική πτυχή του θέματος και έχουμε και ένα πρόγραμμα για πρώτη φορά που είναι πρόγραμμα μακροχρόνιας κατάρτισης της Σεχέλες για τους νέους ακτοφύλακες. Είναι για 27 εβδομάδες. Άρχισε στην αρχή αυτή της χρονιάς και είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα τόσο μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σίγουρα θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις εχέλες και για την αποστολή μας. Αναπτύξαμε επίσης και προγράμματα κατάρτισης διδασκόντων. Το κάναμε στις εχέλες και έχουμε αρχίσει να δίνουμε και εξοπλισμό, όπως σας είπα, σε αυτές τις δύο χώρες, για τις οποίες ο αντίκτυπος της αποστολής μας είναι ήδη ορατός. Οι Σεχέλες καλύπτουν ένα τεράστιο γεωγραφικό χώρο. Έχει κάτω από 5.000 κατοίκους, αλλά το... η επιφάνεια που καλύπτει είναι όση και της Ουκρανίας. Καταλαβαίνετε δηλαδή για τι πράγμα μιλάμε. Γιατί μέγεθος μιλάμε, οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι και η πρόκληση που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα. Σεχέλες και Τζιμπουτή λοιπόν, εκεί έχουμε ήδη ορατά αποτελέσματα και επιτυχίες. Στη συνέχεια, στην Τανζανία, στην αρχή είχαμε δυσκολίες, γιατί οι κάτοικοι εκεί δεν βλέπαν το ενδιαφέρον να έχουν μια τέτοια αποστολή. Οι εξελίξεις όμως ήταν θετικές και αρχίσαμε και εκεί οι δραστηριότητες από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς με ένα πρόγραμμα κατάρτισης για την ε, αστυνομία της θάλασσας και γενικότερα την αστυνομία της χώρας για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Στην Κένια δυστυχώ τα πράγματα είναι λιγότερο καλά. Γιατί ναι, μεν πήραμε ένα γενικό γράμμα που μα καλούσε εκεί, τελικά όμω με την Κένια δεν μπορέσαμε ποτέ πραγματικά να αρχίσουμε μια συνεργασία. Ερχόμαστε τώρα στην καρδιά τη αποστολή μα, που είναι βέβαια η Σομαλία. Είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, γιατί ακριβώ εκεί είναι που η ασφάλεια είναι η πιο δύσκολη. Και μάλιστα χειροτερεύει στο Μογκαντήσιο ιδιαίτερα κάτι που δεν μας διευκολύνει τη ζωή. Η στρατηγική που ακολούθησε η αποστολή UCAP Nestor στη Σομαλία είναι δυτή. Συνεργαζόμαστε με την κεντρική κυβέρνηση με την οποία έχουμε καθημερινά σχέσεις. Υπάρχει ένας σύμβουλος του ναυτικού που είναι στο Μογκαντήσου περίπου βημονή μου βάσεως και συνεργάζεται με τις κεντρικές αρχές της χώρας. Συγχρόνως όμως εκ παραλίλου προσπαθούμε να έχουμε επαφές στις διάφορες περιφέρειες. Γιατί όντως οι περιφέρειες είναι εκείνες που στην πραγματικότητα έχουν την ευθύνη του θαλάσσιου χώρου. Συνεπώς, αναπτύξαμε αυτή την παράλληλη στρατηγική, δηλαδή ενημερώνουμε την κεντρική ε, δίκηση, υπάρχει πλήρης διαφάνεια, αλλά συγχρόνως συνεργαζόμαστε άμεσα με τις περιφερειακές αρχές και ιδιαίτερα με το Πούντλαντ που έχει μια αρκετά αναπτυγμένη διοικητική δομή και τη Σομάλιλαντ. Με τη Σομάλιλαντ είναι ένα καλό παράδειγμα. Εκεί στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς είχαμε μια συνάντηση. Χρησιμοποίησαμε τα μέσα της Αταλάντης. Να, εδώ είναι που συνεργαζόμαστε με την Αταλάντη στενά. Σε ένα σκάφος της Αταλάντης λοιπόν καλέσαμε τις αρχές της Σομάλιλαντ προκειμένου να συζητήσουμε για τη μελλοντική συνεργασία. Ήταν πολύ θετική η επαφή αυτή. Φτιάξαμε έναν χάρτη πορείας με το Somaliland και ετοιμάσαμε στη Αγγίσα, έχουμε ένα γραφείο ήδη και από το γραφείο αυτό και με μέσα ασφάλειας που έχουμε εκεί μπορούμε καθημερινά να συνεργαζόμαστε με τις αρχές της Somaliland που έχουν βέβαια ακτοφυλακή που χρειάζεται όμως κατάρτιση και δουλεύουμε και πάνω στο νομικό πλαίσιο γιατί μας ζήτησαν να τους βοηθήσουμε να συντάξουν νομοθεσία για τον έλεγχο του θαλάσσιου χώρου και των ακτών. Άρα η δουλειά μας εκεί είναι καθημερινή και αποτελεί ένα παράδειγμα για ολόκληρη τη Σομαλία. Προσπαθούμε τώρα να κάνουμε το ίδιο με το Πούντλαντ. Την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα οργανώσαμε μια συνάντηση που την γίδα της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σομαλία στα νυχτά του Μποσάσο με τον πρόεδρο Αντιουίλη και τους περισσότερους υπουργούς. Το θέμα της θαλάσσιας ασφάλειας ήταν βέβαια στην καρδιά της συζήτησης και η Γιούκα Πνέστορ πρότεινε και εκεί ένα χάρτη πορείας προκειμένου να καταρτιστούν οι δυνάμεις της περιοχής και όπως και με τη Σόμιλαντ να έχουμε κάποιους ομολόγους, να υπάρχει μια διοικητική δομή παρόλο που είναι πιο αδύναμη στο Πούτλαντ. Παρ' όλα αυτά εντοπίσαμε κάποιες δυνατότητες. Και άρχισε και η συνεργασία με το Πούντλαντ. Αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής είναι ότι πολύ σύντομα θα καταρτήσουμε στο Τζιμπουτί, είπαμε στο Τζιμπουτί για λόγους ασφάλειας, 30 μέλη των αστυνομικών δυνάμεων του Μποσάζο, που είναι λιμενικές αρχές ουσιαστικά. Θα τους καταρτήσουμε για 6 εβδομάδες στο Τζιμπουτί, μαζί με 20 μέλη της ακτοφυλακής του Μοτάγκου, που είναι το κρατήριο που βρίσκεται κάτω από το Πούντλαντ και όπου η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη ακόμα. Γιατί και εκεί είναι συζητήσιμη η κατάσταση. Συνεπώς θα έχουμε την κατάρτιση αυτή από μέσα Απριλίου μέχρι μέσα Μαΐου στο Τζιμπουτί. Να λοιπόν ένα σημαντικό δείγμα της δράσης της ε, UCAP Nestor στο Πούντλαντ και αλλού. Στο Σομάλιλαντ είπαμε συνεργαζόμαστε με τις περιφερειακές αρχές και σύμφωνα με τη στρατηγική που σας περιέγραψα πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην καρδιά της περατείας που είναι συνήθως στο Πούντλαντ και στο Καλιμούντο. Έτσι λοιπόν, τι θα γίνει στη συνέχεια. Θα υπάρξει μια αναθεώρηση της στρατηγικής όπως ακούσαμε βάσει των εντολών που παίρνουμε από τα κράτη-μέλη που μας λένε να επικεντρωθούμε ακόμα περισσότερο τώρα από ό,τι στο παρελθόν στη Σομαλία. Ήταν ένα σαφές μήνυμα που έστειλαν οι χώρες μέλη να κάνουμε περισσότερα στη Σομαλία μας είπαν. και ιδιαίτερα στο Πούντλο και το Μαγκμπού. Θα υποφεληθούμε λοιπόν από την επιτυχία που έχουμε μέχρι τώρα στην περιφέρεια, ώστε τα δύο επόμενα χρόνια να επικεντρωθούμε περισσότερο στις δύο αυτές υποπεριφέρειες. Το μέλλον είναι βέβαια και η Ιεμένη, γιατί στην Ιεμένη θα αναπτύξουμε και εκεί έναν αξιωματούχο όπου να είναι. Μας ζήτησαν την UCAP Nestor δηλαδή και πήγαμε πρόσφατα στη Σάνα και συζητήσαμε για να δούμε τι μπορεί να καλύψει η UCAP Nestor. Σιγά σιγά λοιπόν θα ανταποκριθούμε στο αίτημα. Η κατάσταση είναι βέβαια δύσκολη, γι' αυτό σιγά σιγά θα προχωρήσουμε στην Ιεμένη. Πάντως μας υποδέχτηκαν οι αρχές πολύ θετικά. Τις επόμενες εβδομάδες λοιπόν θα έχουμε εκεί έναν αξιωματούχο σύνδεσης και στην Ιεμένη. Να σας πω και δύο λόγια τώρα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Η πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι το θέμα της ασφάλειας βέβαια, κυρίως στο Μογκαντούσου. Η κατάσταση δυστυχώς δεν βελτιώνεται. Για να βγούμε λοιπόν ήδη από το αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο δεν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόσβαση, υπάρχει ασφάλεια ικανοποιητική. Αλλά για να βγει κανείς από το αεροδρόμιο, σήμερα δυστυχώς είναι πολύ περίπλοκο. Και η κατάσταση μάλιστα θα έλεγα ότι σήμερα είναι χειρότερη από ό,τι ήταν πριν από ένα-δύο χρόνια. Σήμερα δεν έχουμε τα μέσα εξαιτία αυτή τη δυσκολία τη ασφάλεια, δεν έχουμε τη δυνατότητα να συμβουλεύσουμε τι αρχέ τη Ομαλία, να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή μα δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε να στείλουμε έναν σύμβουλο στη Σομαλία εκεί όπου εδρεύουν οι αρχές της χώρας, εξαιτία του προβλήματος της ασφάλειας, που είναι το κυριότερο πρόβλημά μας. Στο Μογκαντούσου κυρίως, όχι στην Κέσα, Γι' αυτό και επικεντρώσαμε στη Σομάλιλαντ τις προσπαθίες μας. Εκεί η ασφάλεια είναι καλύτερη. Δεν λέω ότι είναι τέλεια, αλλά είναι καλύτερη. Και μπορούμε εκεί να δουλέψουμε. Η δεύτερη δυσκολία μας είναι η πολιτική αστάθεια στην κεντρική δίκηση της Σομαλίας. Κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα ο διάλογος που έχουμε αρχίσει τις τελευταίες εβδομάδες δεν έχει καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο πλήρες σχέδιο που να μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με την κεντρική δίκηση σε ένα σαφέστερο νομικό πλαίσιο. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τι ακριβώς θέλει η κεντρική κυβέρνηση της Σομαλίας για να ελέγξει το θαλάσσιο χώρο της. Για παράδειγμα, δεν έχουν ε, ε, δηλώσει ποια είναι η αποκλειστική οικονομική του ζώνη. Γιατί αν θέλει κανείς να ελέγξει ένα χώρο, πρέπει να ξέρει ποιο είναι ο χώρο αυτό, να οριοθετήσει το χώρο που θέλει να ελέγξει. Δεν έχει γίνει όμω αυτό ακόμα. Συνεπώ, για να ολοκληρώσω, Πρόεδρε, θα έλεγα ότι η πειρατεία είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η ρύθμιση τη δραστηριότητα στη θάλασσα τη πειρατεία, και αυτό το κάνει πάρα πολύ καλά η Αταλάντη και όλο και καλύτερα μάλιστα. Το δεύτερο επίπεδο είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων ελέγχου των ακτών, η UKAP το κάνει αυτό. Βέβαια η απάντησή μας είναι μερική προς το παρόν. Και το τρίτο, το πιο δύσκολο, είναι να δώσουμε δραστηριότητες, οικονομικές αναλλακτικές δραστηριότητες, στους ανθρώπους που ζουν στις ακτές και οι οποίοι έχουν στραφεί στην πειρατεία γιατί δεν βλέπουν να έχουν άλλες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης εκεί που ζουν. Αυτό βέβαια είναι περισσότερο αποστολή αναπτυξιακή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τόσο τη UCAP Nestor, αλλά αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Γιατί οι συνομιλητέ μα εκεί μα λένε ότι όσο δεν έχει διακανονιστεί και το θέμα αυτό τη ανάπτυξη τη Σομαλίας, των ακτών τη χώρα δηλαδή, το φαινόμενο τη πειρατεία θα παραμείνει και κάθε φορά που θα υπάρχει ευκαιρία οι άνθρωποι εφόσον δεν θα τους φτάνει η αλεία ή δεν έχουν τέλο πάντων άλλες δραστηριότητες θα στρέφονται πάντα στην πειρατεία. Και για να το δούμε αλλιώς υπάρχουν... Ε, υπάρχει θεραπεία που θα έλεγα ότι είναι, ή ε, μάλλον υπάρχει παρηγοριά θα έλεγα που είναι η Αταλάντη, υπάρχει η θεραπεία που είμαστε εμείς, η Γιου και υπάρχει και η πρόληψη που είναι η ανάπτυξη της Σομαλίας. Άρα η παρηγορητική, η θεραπεία και η πρόληψη. Θα τα έλεγα και έτσι αυτά τα τρία επίπεδα. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι ερωτήσεις έχετε. Σας ευχαριστούμε για αυτή την τόσο πλήρη παρουσίαση. Πριν να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, έχω μία ερώτηση που αφορά τους άλλους ε, διεθνούς ε, φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στην πολιτική που διεξάγεται στην περιοχή. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υπάρχουν, το Μάρσικ, το Μάζε και καλύπτουν και την ε, θαλάσσια εποπτεία. Υπάρχουν προγράμματα που δεν θα πω ότι είναι ανταγωνιστικά, αλλά διμερεί ή από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτες χώρες, ιδιαίτερα σκέφτομαι τις ΗΠΑ. Υπάρχουν δηλαδή προγράμματα που υπάρχουν και θα μπορούσαν να λειτουργούν αν θέλετε στην ίδια σφαίρα στην οποία κινείστε κι εσείς. Επίσης, ο κύριος Γκάλερ θέλει να πάρει το λόγο, τον δίνω μέσος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για τη διάλεξη. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε και επίσης και για αυτή τη μεγάλη απλωμένη βεντάλια δραστηριοτήτων αλλά και συνεργασίας που μας ε, παρουσιάσατε ανάμεσα στις ε, διάφορες αποστολές ε, που έχουμε επιτόπου. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλό που είμαστε παρόντες, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα, όπως είπατε κι εσείς, ε, εάν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με την κυβέρνηση της Σομαλίας ως προς τους ε, στόχους της, δηλαδή θα θέλαμε να υπάρχει μια ισχυρότερη βάση συνεργασίας ε, για να μπορούμε να προβάλλουμε καλύτερα τη στρατηγική μας. Από ό,τι λοιπόν ε, γνωρίζω, για αυτές τις παράλληλες αποστολές για το 2012 έχει, ε, από το 2012 έχει δραστηριοποιηθεί και το επιχειρησιακό μας κέντρο, από ό,τι εξ όσων γνωρίζω. Ακούω βέβαια ότι η λειτουργία ενός τέτοιου επιχειρησιακού κέντρου που είναι να συντονίζει τις δραστηριότητες για να υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα. Από ό,τι φαίνεται αυτό το επιχειρησιακό κέντρο δεν μπορεί να εκπληρώσει την επιστολή του γιατί τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουν και ορισμένοι λένε στο τέλος αυτό το επιχειρησιακό κέντρο δεν προσφέρει καμία υπεραξία και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ λυπηρό, γιατί εγώ θέλω να κάνουμε πράγματα που προσφέρουν υπεραξία. Μήπως μπορείτε λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας, τι ακριβώς ε, διαδραματίζεται και αν τελικά πράγματι αυτό το κέντρο δεν είναι αποτελεσματικό, τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Ίσως την ε, απάντηση θα μπορούσε να τη δώσει ο κύριος Ζανβιέν και βγαίνουμε λίγο από το θέμα μας. Ο κύριος Βανόρτ. Um, Πολύ ενδιαφέρουσα η διάλεξή σας, η ομιλία σας, αλλά νομίζω ότι τελικά ε, μας άφησε περισσότερα ερωτήματα από αυτά που είχαμε πριν από την ομιλία σας. Ε, η κατάσταση όσο εξελίσσεται τα τελευταία δύο χρόνια θα μας ενδιαφέρει να ακούσουμε πόσα κονδύλια έχουν δαπανηθεί για αυτή την κατάσταση και ποια είναι η υπεραξία που επιτύχαμε. Και θέλω να πω, όταν μιλάμε για την ε, αντιμετώπιση της πειρατεία. Κουράστηκα να ακούω για αυτά που υποτίθεται ότι πέτυχε η αποστολή Αταλάντη. Κάθε άλλο τελικά το μόνο που ήταν αποτελεσματικό ήταν το μισθωμένο ένοπλο προσωπικό πάνω στα πλοία. Αυτό έκανε τη διαφορά στον Ινδικό ωκεανό και στο κέρας της Αφρικής ε, στις ε, χώρες που αναφέρατε. Όχι ότι θέλω να πω ότι δεν ε, προσέφεραν τίποτα οι θαλάσσιες περιπολίες ε, των ε, κρατών μας. Αλλά και εδώ πάλι βλέπουμε άλλο ένα παράδειγμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να παίξει κάποιο ρόλο, ε, ανταποκρίνεται σε εκκλήσεις και διερωτώμε τελικά το κατά πόσον αυτές οι προσφορές που κάνατε, κατά πόσον θα γίνουν αποδεκτές ή όχι. Νομίζω όλο αυτό είναι πολύ αμφιλεγόμενο και το θέμα είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσον όλα αυτά είναι αποδεκτά, αν είναι η σωστή απάντηση. Εξάλλου υπάρχει και μία σχέση ανάμεσα σε αυτό που λέτε εσείς και την ευρύτερη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά μας ανησυχούν ιδιαίτερα και βεβαίως ε, δεν σχετίζονται επουδενή με το ρόλο άλλων οργανώσεων όπως είναι προπάντων το ΝΑΤΟ. Όπως ξέρετε το ΝΑΤΟ έχει τη δική του θαλάσσια στρατηγική τις συμμαχίας και αυτό δεν αναφέρεται σχεδόν πουθενά στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξετάζουν την κατάσταση. Και επίσης δεν αναφερθήκατε και στην Αφρικανική Ένωση, στο ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει ε, πιο έντονο ρόλο αυτή, αυτός ο φορέας. Εάν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να βοηθήσει υπάρχουν ένα-δύο πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν που όμως δεν έχουν σχέση με αυτή την υποτιθέμενη αμυντική πολιτική στην οποία θέλουν να εντάξουν τα πάντα. Ας δούμε παραδείγματος χάνει το θέμα της πειρατείας και τα χρήματα που συνδέονται με αυτήν. Η δουλειά που γίνεται για να εντοπιστούν οι διεθνείς διασυνδέσεις της ε, πειρατείας, οικονομικές διασυνδέσεις, αυτό ήταν πολύ πολύ και εκεί ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει περισσότερα. Όσον αφορά την επιβολή νομικών δομών, ε, μια υποδομή νομική σε χώρε όπω η Σομαλία, δεν ξέρω, έχω επιφυλάξει γιατί τελικά ε, θα υπάρξει μια ε, γραφειοκρατία νομική που ταιριάζει περισσότερο σε δυτικέ χώρε και όχι για αυτή για την οποία μιλάμε και παρεμπιπτόν σα συστήνω επιφύλακτα την ταινία Captain Phillips γιατί παρότι είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας παρόλα αυτά εκεί ε, έχει πολλά και καλά μαθήματα και το μεγαλύτερο μάθημα που εξάγει κανείς είναι ότι μια σωστή πράξη από την αρχή θα μπορούσε να βάλει τέλος ε, σε αυτό που προέκυψε στην ταινία ε, και στην ε, ενέργειες που ακολούθησαν και που ε, στήχησαν εκατομμύρια. Με μία λίρα θα μπορούσε κανείς να λύσει το πρόβλημα της εξαρχής, αλλά εντάξει, αν γινόταν αυτό, τότε υπήρχε εκεί ταινία. Ποιο θα ήταν το σενάριο της ταινία. Δεν ξέρω ποιος θέλει να απαντήσει. Ο κύριος Ζανβιέ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι και κύριοι βουλευτέ, θα επικεντρώσω τι απαντήσει μου στην υποστήριξη που παρέχουμε στα πλαίσια αυτού του επιχειρησιακού κέντρου με την δομή των Βρυξελών. Πρόκειται για μια δομή που δημιουργήθηκε εδώ και δύο χρόνια. Η διοίκηση της άρχισε τώρα πρόσφατα και διαθέτουμε τις ε, δομές για την διαχείριση των κρίσεων στρατιωτικών και μη για να βελτιώσουμε τον συντονισμό όλων των συνιστοσών έτσι όπως ε, τις περιέγραψε την εισαγωγή του παρατήρηση ο πρόεδρος, την Ιντεάντε, την δράση για τη Σομαλία και την UCAP Νέστορ, την αποστολή αυτή που δημιουργήθηκε το 2012. Πρόκειται για ένα μέσο ad το οποίο έχει αναλάβει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το συντηνιστικό ρόλο και διευκολύνει την δράση των τριών αποστολών και όλων των άλλων δομών που ανέφερε ο πρόεδρος με την ε, συνδρομή της Επιτροπής που είναι το μέσον που μας επιτρέπει να αναπτύξουμε όλα τα μέσα που έχουμε ώστε να έχουμε στοχευμένη προσέγγιση στα θέματα που υπάρχουν όχι μόνο για να καταπολεμήσουμε την ε, πειραντία αλλά μακροπρόθεσμα όπως είπε και ο ε, σε Ετιέν για να ακολουθήσουμε μια σωστή πολιτική. Όπως κάθε νέο μέσον, δεδομένου ότι το κέντρο διαχείρισης αυτό δημιουργήθηκε εκτός της δομής της ε, ε, στρατιωτικής κεντρικής ένταση την οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέσον αυτό έχει μία αποστολή ιδιάζουσα, ad hoc. και χρησιμοποιεί συστήματα που έχουν οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσματα. Ανταποκρίθηκε για το μη στρατιωτικό σκέλος σε όλες τις προσδοκίες και αποτελεί και την διεπαφή μεταξύ της Επιτροπής, στην οποία υπάρχουν οι εξωματικοί σύνδεση και του πυρήνα για την διαχείριση κρίσεως της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, χωρίς να πω σε λεπτομέρειες, σε σχέση με τις παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν από τους αξιότιμους ε, βουλευτές και κυρίως των βουλευτής της Μεγάλης Βρετανίας, ήθελα να σας πω ότι εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, των δράσεων του ΝΑΤΟ και της Αφρικανικής Ένωσης, εάν αυτό δεν αναφέρεται στην εισαγωγική παρατήρησή μου, δεν το έκανα διότι δεν νομίζω ότι δεν είναι χρήσιμες, αντιθέτως, απλώς θέλησα να εστιάσω την προσοχή μου στην αποστολή αυτή που είναι μη στρατιωτική και να σας εξηγήσω ποιο είναι το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η αποστολή Ιού Καπνέστορ. Φαίνεται ότι θα μπορούσε να αναθεωρηθεί ο στόχο της αποστολής μας και δεν ανέφερα ότι είμαστε και σε στενή συνεργασία και σχέση με τους άλλους φορείς της Europol και των Ηνωμένων Εθνών που αναπτύσσονται, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά τα μέσα ε, που χρησιμοποιούνται οι ε, οικονομικές ε, παράνομες δραστηριότητες, της ε, πειρατείας και όλα αυτά μπορούν να περιχαρακωθούν και να βεβαιωθούμε ότι όλα γίνονται με νόμιμο τρόπο. Επίσης, κρίνουμε ότι ο σύνδεσμος που θα έχουμε με την ε, ε, η εμένη θα είναι χρήσιμες εξαιτίας της μεταφοράς κονδυλίων και της ανάπτυξης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων που ενδεχομένως θα αναπτυχθούν σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Euh, Ευχαριστώ. Θέλω να συμπληρώσω και εγώ λιγάκι το θέμα των διεθνών παραγόντων που δρούν και εμείς συνεργαζόμαστε μαζί τους για την καταπολέμηση της πειρατείας. Θα έλεγα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που δρούν στο κέρας της Αφρικής και σίγουρα χρειάζεται καλός συντονισμός. Αυτό όμω δείχνει πόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχει η διεθνή κοινότητα για την περιοχή αυτή προκειμένου να αντιμετωπίσει την μάστιγα αυτή τη πειρατεία αποτελεσματικά. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν δύο μέσα. Υπάρχει το ΜΑΣΕ και το ΜΑΣΕΚ, δύο προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καλύπτουν τον εξοπλισμό και την ενίσχυση δυνατοτήτων στην περιοχή. Έχουμε λοιπόν σχέσεις με τα δύο αυτά προγράμματα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και να έχουμε έναν συντονισμό μεταξύ μας, να προχωρήσουμε και στον εξοπλισμό με σκάφη ή άλλου είδους εξοπλισμό. Δουλεύουμε λοιπόν πάνω σε αυτά και από αυτόν έχουμε και τη στήριξη του ΟΨΕΝ που αναφέρθηκε από σας Ως αποστολή εποφεληθήκαμε από τη στήριξη του Όψεν λοιπόν για να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερο συντονισμό με τα προγράμματα αυτά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, υπάρχει και η ΓΕΤΕΣΕ που δρά όσον αφορά την πειρατεία. Για παράδειγμα, φτιάχνει τις φυλακές, γιατί άπαξ και δικαστούν οι πειρατές εγκλείονται σε φυλακές βέβαια. Δεν αποτελεί μέρο βέβαια τη εντολή μας. Εμείς από τη στιγμή που ο πειρατή καταδικάζεται ή φέρεται στη δικαιοσύνη, σταματούμε. Δεν ασχολούμεθα με την εκτέλεση της ποινή. Αυτό είναι κάτι που το κάνουν οι υπόλοιποι. Με κοινωτικά κονδύλια μάλιστα. Συνεργαζόμαστε, είπαμε, με την Somaliland, με το UNDC, προκειμένου να υπάρχει καλός καταμερισμός και να μην υπάρχει επικάλυψη. Είναι καθημερινή η επαφή που έχουμε επίσης με τα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα όσον αφορά ε, διμερός, συνεργαζόμαστε με την Τουρκία, η οποία έχει πρόγραμμα στήριξης του ναυτικού της Ομαλίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης διμερές πρόγραμμα με τη Σομάλιλαντ. Η Ιαπωνία έχει επίσης συνεργασία με την ακτοφυλακή του Τσιμπουτή. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επίσης δικές τους δραστηριότητες. Άρα ναι, φυσικά και υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που δρούν στην περιοχή και ο συντονισμός είναι ένα ζήτημα. Όλοι όμως πάμε προς την ίδια κατεύθυνση και αποφεύγουμε τις επικαλύψεις. Και όσο πιο πολύ τις αποφεύγουμε, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε όλοι μαζί, αντί ο καθένας μόνος του. Μέρος της δουλειάς μας είναι ακριβώς η συμμετοχή μας σε ομάδες συντονισμού. Πολλές από αυτές τις συναντήσεις γίνονται στον αερόμπι. Πρόεδρος, καλώς. Δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ε, θέλω να σας υπενθυμίσω λιγάκι αυτό που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει το Q-Cup Store Nestor και υπάρχει και για τα Λάντι. Αυτά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Είναι αλήθεια ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ οι δραστηριότητες των πυρετών. Αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό πράγματι στο γεγονός ότι υπάρχουν ένοπλοι πάνω στα σκάφη. παρόλα αυτά υπάρχει και μια δύναμη αποτροπής εξαιτία των σκαφών που βρίσκονται στη θάλασσα. Η ενημέρωση, η χαρτογράφηση του φαινομένου με ε, ελέγχους από αέρος είναι επίσης κάτι αποτρεπτικό. Άρα θα έλεγα ότι είναι πολύ βιαστικό να λέμε ότι μειώθηκε η πειρατεία εξαιτία του ενό ή του άλλου παράγοντα. Γιατί οι διάφοροι παράγοντες οι αποτρεπτικοί μεταξύ τους συμπληρώνονται. Έτσι καλώς υπάρχει η ανάγκη για πολύ προσοχή μας. Το λένε οι άνθρωποι επιτόπου γιατί δυστυχώς το φαινόμενο μετακινείται πάρα πολύ γρήγορα. Συνεπώς άπαξ και υπάρξει κάποια δυναμία κάπου θα αποφεληθούν οι πειρατές και θα δραστηριοποιηθούν εκεί. Αυτό το οποίο μας εξέπληξε στο Τζιμπουτί ιδιαίτερα είναι το αυξανόμενο ενδιαφέρον και μαζικό θα έλεγα πολλών διεθνών φορέων για την περιοχή και όχι μόνο εξαιτία της πειρατείας αλλά ενδιαφέρονται και για την ε, ανάπτυξη της περιοχής και για τις στρατιωτικές ε, δραστηριότητες. Επισκεφθήκαμε λοιπόν αμερικανικές εγκαταστάσεις, μεγάλες, που επεκτείνονται στο Τζιμπουτί. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλη παρουσία της Ιαπωνίας στο Τζιμπουτί. Οι αρχές του Τζιμπουτί επίσης μας επιβεβαίωσαν ότι οι Κινέζοι και οι Ρώσοι ενδιαφέρονται για στρατιωτικές ναυτικές εγκαταστάσεις. Και η Τουρκία βεβαίως δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν υπάρχει μεγάλη ζήτηση για το Τζιμπουτί. Προκειμένου να υπάρχει εκεί παρουσία διαφόρων πλευρών. Προς το παρόν Υπάρχει η παραδοσιακή παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γαλλίας πιο συγκεκριμένα, η οποία όμως μειώνεται. Και εδώ καλά θα κάνουμε να αναρωτηθούμε. Γιατί τόσοι πολλοί στον κόσμο ενδιαφέρονται για το κέρας της Αφρικής και κυρίως για τον Τζιμπουτί. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο τμήμα του ταξιδιού μας στην Αιθιοπία και την Αφρικανική Ένωση. Οι σχέσεις είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντικές, πολύ έντονες. Δεν είναι πάντα εύκολες, ιδίω με την Αφρικανική Ένωση, γιατί ε, πρέπει να δείχνουμε βαστιτοποίηση η Αφρικανική Ένωση, να, για την Κεντρική Αφρική για παράδειγμα, μας πέρασε το μήνυμα που έλεγε ότι καλό είναι να έχουμε περισσότερο συντονισμό στην αρχή των διαδικασιών. Αν υπάρξει στρατιωτική ευρωπαϊκή αποστολή στην Κεντρική Αφρική, που είναι σε καλό δρόμο από ό,τι έχω καταλάβει σήμερα. Πάντως υπάρχει σύγκληση απόψεων για τη Σομαλία καταρχήν και για τον σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως τον οικονομικό, με μέσα τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη, στην ειρήνη και την ασφάλεια. Αναμφίβολα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος εταίρος της Αφρικανικής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καλλιεργήσουμε περισσότερο, να το διατηρήσουμε και να το υπογραμμίζουμε. Για την Αιθιοπία τώρα. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσε επαφές με τον επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων εκεί, τον Υπουργό Εξωτερικών, Απευθεία επαφές. Δεν μα έκρυψαν ότι υπάρχει κάποιος σκεπτικισμός ή μάλλον αν όχι σκεπτικισμός όσον αφορά την αποστολή Αμισόμ. Η Αιθιοπία εδώ και λίγο καιρό επίσημα συμμετέχει. Συγχρόνως όμως η Αιθιοπία πιστεύει ότι η συντονισμένη λειτουργία δεν είναι αρκετά ικανοποιητική και ότι θα έπρεπε να στηριχτούμε περισσότερο σε διμερείς δράσεις για να, υπάρχουν, να υπάρχει αντίκτυπος. Υπάρχουν επιθέσεις που γίνονται από κοινού με το τσιμπουτί και βοήθεια στην κατάρτιση. Εδώ θα μπορούσαμε να είμαστε πιο επικριτικοί σε αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κατά τη γνώμη τους φαίνεται ιδιαίτερα μετροπαθής και κάπως μακριά από την πραγματικότητα επιτόπου. Πιστεύουν ότι πρέπει να γίνεται κατάρτιση στο έδαφος της Σομαλίας, παρόλο που υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας και αυτό βέβαια αποδυναμώνει κατά πολύ οποιαδήποτε αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως οι επαφές ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Διαπιστώσαμε και την προτεραιότητα που δίνουν οι αρχές της Αιθιοπίας στην κρίση στο Σουδάν. Η Αιθιοπία έχει διαμεσολαβητικό ρόλο εκεί. Η κρίση αυτή, πέρα από την σουδανική πτυχή, αφήνει να διαφανούν οι διαφορές με την Ερυθρέα και την Αιθιοπία. Γι' αυτό και προσέξαμε και εμείς το ρόλο της Ερυθρέας. Μπορεί να γίνεται κάποια υπερβολή όσον αφορά για τον ρόλο αυτό της Ερυθρέας ως κακός μαθητής, αλλά σίγουρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία από τον Τζιμπουτί και από την Αιθιοπία και από την Αφρικανική Ένωση για το πώς να συμπεριφερθούν απέναντι στην Ερυθρία που λένε στην Αιθιοπία ότι αποσταθεροποιούν την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν. χωρίς βέβαια να μπορούμε να πούμε ότι μας δίνουν και αποδείξεις οι Αιθίωπες. Σίγουρα υπάρχουν μεγάλες υπόνοιες για τον ρόλο της Ερυθρέας. Οι εντάσεις, άρα λοιπόν αναζωογονούνται άμεσα στην Ερυθρέα και την Αιθιοπία. Και η Αιθιοπία ακριβώ αυτό που μας είπε είναι ότι η ανησυχία είναι μεγάλη. Καλό λοιπόν θα ήταν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί μήπως υπάρξει νέα κρίση μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Και τέλος, το τελευταίο που μας είπαν οι Αιθίωπες ήταν το θέμα του Νείλου. Και εδώ πολύ δύσκολη κατάσταση με την Αίγυπτο αυτή τη φορά. Και είπαν ότι θα πρέπει να βρεθούν συνομιλητές, τρίτοι συνομιλητές, δεν μίλησαν βέβαια επίσημα για διαμεσολαβητές, αλλά να υπάρξει κάποιος τρίτος συνομιλητής που να βοηθήσει σε κάποια προσέγγιση απόψεων. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει πλήρες αδιέξοδο στο διάλογο μεταξύ της Αιθιοπίας και της Αιγύπτου. Το Νότιο Σουδάν μια φορά παίζει καταλητικό ρόλο. Ο Νείλος όμως προστίθεται και έτσι παραμένει ένα κλίμα ιδιαίτερη δυσπιστία ανάμεσα στην Αιθιοπία και την Αίγυπτο, που είναι στο κάτω-κάτω δύο μεγάλε χώρε στην περιοχή. Στο διευρυμένο κέρα τη Αφρική θα έλεγα. Αυτή ήταν η παρουσίαση. Θα έπρεπε να είχαμε και μια πτυχή για τη Σομαλία αυτή καθ' αυτή και αυτό να το κρατήσουμε γιατί παρά τις δυσκολίες που μας υπογραμμίσατε και ο ένας και ο άλλος για τις δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων στο Μογκαντήσου, παρόλα αυτά εκεί παίζεται το παιχνίδι. Και η Αιθιοπία αυτό ακριβώ μας αποσαφήνισε ότι επιτόπου στη Σομαλία πρέπει να βρεθούν και οι συνομιλητές και οι πηγές για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, χωρίς βέβαια να έχει κανείς υπερβολικές ψευδεστήσεις. Αυτά θα κλείσουμε λοιπόν αυτό το τμήμα της ημερήσιας διάταξης αυτή τη συζήτηση και σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Ο Κρίστοφ Λίζεκ τώρα, ο αντιπρόεδρος μας που ήταν μαζί μας την προηγούμενη εβδομάδα στην Αφρική, θα πάρει τώρα το λόγο για να μας ενημερώσει για την αμυντική βιομηχανία. Μετά από δύο λεπτά διακοπή. Okay, ladies and gentlemen, let's start without any delay. Um, the next steps in strengthening the European defense industry. We have an exchange of view with Mr. Sławomir Tok. Θα μιλήσει τώρα ο κύριος Τοκάρτσκι που το θέμα του είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένα και είναι μια έκθεση που συντάχθηκε τους τελευταίους μήνες από τον κύριο Γκάλα και είχαμε και ε, σχετική ακρόαση ή ακροάσεις. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Τοκάρσκι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που δεν είναι εδώ ο διευθυντής μου αλλά δεν είναι εδώ, έχει να κάνει κάτι που έχει σχέση με το Κοπέρνικους. Να σε εξηγήσω πού ακριβώς ε, βρισκόμαστε μετά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και μετά νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε τις ερωταπαντήσεις. Όπως ενδεχομένως τα ε, γνωρίζετε, από το Δεκέμβρη του περασμένου έτους η αξιολόγηση των συμπερασμάτων ήταν πολύ θετική γιατί ε, οι προτεραιότητες μας στηρίχτηκαν από τα κράτη-μέλη και αποκομίσαμε την εντύπωση ότι πρόκειψε κάτι πολύ σημαντικό στον τρόπο με τον οποίο εξτάζουν τα κράτη-μέλη το όλο θέμα και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, προσέφεραν ε, ενθάρρυνση, κίνητρα για τη δουλειά μας. Μετά λοιπόν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου είχαμε ε, την συνάντηση των Υπουργών Άμυνας στην Ελλάδα και εκεί πάλι στηρίχθηκε το δικό μας το ανακοινωτέν και οι δράσεις μας και είχαμε και μία συνάντηση με την με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας πριν από λίγες μόνο ημέρες ε, και πρέπει να σας πω διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αλλαγή στάσης ανάμεσα στα κράτη-μέλη ε, σε σχέση με την κατάσταση που υπήρχε πριν από 1,5 χρόνο. Νομίζω τώρα όλοι αναγνωρίζουν περισσότερο το θετικό ρόλο που μπορεί να διαρματίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, επίκειται ή σύντομα πρόκειται να έχουμε κάποια στοιχεία της ανακοίνωσης επιτροπής που θα εφαρμοστούν. Ένα από αυτά είναι η ανακοίνωση για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη ε, στον ε, πολιτικό εναέριο χώρο, η ένταξή του σε αυτό το χώρο θα ξεκινήσει και η δουλειά μας για τις ε, προδιαγραφές. Έχουμε προβλέψει μια εντολή για τις προδιαγραφές που έχουν σχέση με την ναυτική ασφάλεια. Προδιαγραφές που έχουν σχέση με τα δεδομένα έτσι ώστε στο μέλλον να είναι δυνατόν να υπάρχει απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε όλους τους χρήστες θαλάσσιου χώρου. Και αυτό έχει σχέση με αυτά που λέμε στο ανακοινωτέν σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής, πάντα σε σχέση με τις προδιαγραφές. Τώρα λοιπόν το επόμενο βήμα είναι η έγκριση του χάρτη πορείας, ο οποίος ε, θα ενημερώσει, θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο και αυτό θα είναι περισσότερο επιχειρησιακό έγγραφο από το ανακοινωτέν. Θέλουμε το εξής, Θέλουμε να είμαστε πιο επιχειρησιακοί σε σχέση ε, με αυτό που πρωτοπροτείναμε τον Ιούλιο, δηλαδή να εξηγήσουμε ποιες είναι οι λεπτομέρειες αυτών των δράσεων, πώς πρόκειται να αναπτυχθούν και τι είδους ε, στόχους ε, μπορούμε να θεωρούμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε. Και πρέπει να διευκρινιστούν κάποιοι εξ αυτών των στόχων και αυτό έγκαιρα πριν από την επόμενη συζήτηση που θα γίνει ε, στις 15 Ιουλίου. Να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι πραγματικά κάτι προσφέρουμε και ότι μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε και τον πολιτικό ενθουσιασμό που προέκυψε από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Και κάτι άλλο. Το ανακοινωτέν αναφέρεται στο μηχανισμό διαβουλεύσεων ε, με τα κράτη-μέλη. Σε αρκετούς ε, τομείς ε, έχουμε ένα τέτοιο μηχανισμό. Παρήματος χάρη όσον αφορά την τυποποίηση, η δουλειά γίνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Ε, όπως και στην ενέργεια, θα κάνουμε χρήση των ε, ομάδων εμπειρογνωμόνων που υπάρχουν, αλλά θέλουμε επίσης να προσφέρουμε στα κράτη-μέλη την ευκαιρία να προβούν σε αναθεώρηση για να δουν κατά πόσον μπορούν να έχουν πιο σωστή άποψη για την εφαρμογή του συνόλου των δράσεων. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο κάθε κάποιους μήνες ε, θέλουμε να έχουμε μια οριζόντια συνάντηση και αυτή προβλέπεται τώρα να λάβει χώρα στις 14 Μαΐου. Όσον αφορά τώρα την ε, έκθεση, αυτή ε, θα κατεθεί τον Ιούλιο υπό την Ιταλική Προεδρία και από τις πρώτες επαφές που είχαμε με την Ιταλική Προεδρία καταλήξαμε στο ότι την έκθεση αυτή ενδέχεται να τη συζητήσουμε τον Οκτώβριο ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τοκάρσκι. Ο κύριος Γκάλα, ο Μάικλ, ε, Μίκαλ θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω για αυτά που μας ε, είπατε, όπως επίσης και για την ε, ενημέρωση σχετικά με τη δική μου την ε, έκθεση η οποία εγκρίθηκε στις 4 Φεβρουαρίου από την Επιτροπή. Χαίρομαι πάρα πολύ που η έκθεσή μου συνοψίστηκε σε αρκετά σημεία και έχω και κάποιες ερωτήσεις. Εκτός από τη δική σας τη Γενική Διεύθυνση συμμετείχαν και άλλες ε, στην κατάρτιση αυτής της έκθεσης follow-up. Συντονίστηκαν οι Γενικές Διευθύνσεις και αν όχι γιατί όχι. Και κάποια άλλα σημαντικά σημεία της έκθεσης ε, δεν τοποθετηθήκατε επί σημαντικών θεμάτων όπως για το διάστημα και για τον κυβερνοχώρο. Δεν μας είπατε τίποτα γι' αυτά. Στο θέμα των ερευνών δεν προβλέπετε follow-up για την πρόταση μας ε, με βάση το άρθρο 185 που αναφέρεται στη δυνατότητα συγχρηματοδότησης ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ένα άλλο ερώτημα. Στις 4 Μαρτίου η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να δεχτούν αυτό ή πήραν αυτό το χάρτη πορείας. Γιατί λοιπόν αυτό δεν το διαθέσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, ως Κοινοβούλιο είχαμε συμφωνήσει, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ελήφθη απόφαση ότι θα υπάρξουν σε ολόκληρη την Ευρώπη προδιαγραφές ε, έτσι ώστε να υπάρξει εξοικονόμηση των δαπανών κατά την τυποποίηση. Τώρα όμως με ενημέρωσαν ότι ένας από τους οργανισμούς ε, τους ευρωπαϊκούς τυποποίησης απορρίπτει να υπάρχει ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας ε, για τα αμυντικά προϊόντα. Έχετε ενημερωθεί επ' αυτού και τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να μπορεί να αποδίδεται αυτή η ετικέτα ποιότητας από ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Όσον αφορά τώρα στην ε, διάσκεψη που ήμουν και εγώ παρόν, εκεί αναφέρθηκε ότι η Κομισιόν προτίθεται από το 2018 να καταθέσει preparatory action για την έρευνα. Και γιατί τόσο αργά. Στην έκθεσή μου καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ξεκινήσει με το θέμα αυτό ώστε δυνατόν νωρίτερα στο νέο ε, χρηματοδοτικό πλαίσιο. Εάν λοιπόν περιμένουμε ακόμα περισσότερο ε, για να ε, προσελκύσουμε εμπειρογνώμονες από ορισμένους τομείς σε άλλους, τότε νομίζω ότι δεν θα έχουμε πάρα πολλά θέματα για να εξετάσουμε. Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές τα ερωτήματά μου και κυρίως όσον αφορά το θέμα γιατί ε, θα αργήσετε, θα καθυστερήσετε τόσο πολύ με την προκαταρκτική ε, πράξη, preparatory action. Τέλος, παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε. Ευχαριστούμε πολύ, Μάικλ, για αυτές τις τόσο πολλές ερωτήσεις, πολύ σημαντικές βεβαίως. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Κύριε Τοκάρσκι, έχετε το λόγο. Πρόκληση πάντα. Πρόκληση να απαντά κανείς στις ερωτήσεις του Μάικλ το πρώτο ερώτησα που αφορά τις ε, ε, διαβουλεύσεις μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών έχουμε μια ειδική task force και όλες οι δράσεις που έχουν συμπεριληφθεί στην ανακοίνωση έχουν ζητηθεί από task force που έχει δει συναντηθεί, θα και πάλι και είμαστε σε επαφή συνέχεια με τις άλλες διευθύνσεις κυρίως αυτή που αφορά τα θέματα που αφορούν με τις αγορές, αλλά και με τις άλλες γενικές διευθύνσεις που έχουν σχέση ε, ως αρμόδιες με τα θέματα τα οποία χειριζόμαστε. Υπάρχουν λοιπόν διαβουλές σε τακτάς διαστήματα και όπως σας είπα όλες οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχουν όχι διότι αυτή ήταν η ιδέα ε, πίσω από την δημιουργία αυτής της Task Force, αλλά προσπαθούμε να εξετάσουμε οριζοντίως τι μπορεί να κάνει για την αμυντική αυτή πολιτική όλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη στα πλαίσια Τώρα, όσον αφορά το ίντερνετ και τον κυβερνοχώρο, την ανταγωνιστικότητά μας. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν τα σχετικά συμπεράσματα. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι από κοινού να πάρουμε ε, μέτρα για την παρακολούθηση των μέτρων αυτών. Υπάρχει η στρατηγική του και η ασφάλεια του, του κυβερνοχώρου, το οποίο ασχολούνται οι δικές υπηρεσίες της Επιτροπής, εκτός από το πρόγραμμα που έχει σχέση με την ασφάλεια του κυβερνοχώρο στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 υπάρχει και η σχετική οδηγία που αφορά την ε, σύμπραξη του δικού και δημόσιου τομέα για θέματα ασφαλείας. Αυτό ήταν στο πρώτο, πρώτη ομάδα των συμπερασμάτων στα οποία καταλήξαμε, αλλά η παρακολούθηση εκ μέρους της Επιτροπής αφορά και επόμενα στάδια. Στο θέμα του οδικού χάρτη. Αυτό ήταν ένα έγγραφο εργασία που προετοιμάστηκε για την άτυπη ε, συνάντηση υπουργών στην Αθήνα. Πρόκειται για έναν πίνακα με διάφορα στοιχεία για να κατανοήσουν οι πάντες καλύτερα πώς θα μπορούσαμε να συντονιστούμε. Εκτενής κατάλογος 65 δράσαμε. Ποιος είναι υπεύθυνο για κάθε δράση και νομίζω ότι μπορούμε να ζητήσουμε στην γραμματεία του Συμβουλίου να σας στείλει τον κατάλογο αυτό των δράσεων για να ενημερωθείτε. Όλον αφορά την τυποποίηση και την πιστοποίηση. Όπως σας είπα, πρόκειται για δύο τομείς του οποίους υπάρχει πολύ στενή συνεργασία. Στον τομέα της τυποποίησης υπάρχουν δύο σικές ιδέες. Πρώτα απ' όλα να δώσουμε μεγαλύτερη ισχύ στην ομάδα για θέματα πιστοποίησης που δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί ως το σώμα το οποίο συντονίζει ό,τι αφορά την τυποποίηση. Δεύτερη ιδέα να προσφέρει η Επιτροπή στα πλαίσια της ομάδας αυτής για τους κανόνες και τα στάνταρ, τα οποία και τις που χρειάζεται η δική βιομηχανία. Κάτι το οποίο θα πρέπει να περάσει από τους ευρωπαϊκούς ε, οργανισμούς πιστοποίησης και να δούμε μετά τι συγκεκριμένο θέμα θέλουν να προβάλλουν και να λύσουν μέσω αυτής της ομάδας τα κράτη-μέλη. Και όπως σας είπα ήδη, τέθηκε σε εκκίνηση το ρογιαμό εργασία το οποίο ε, πράγμα το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί σε θέματα θαλασσίου χώρου και από του χρόνου για στρατιωτικούς και μη σκοπούς με την παροχή πληροφοριών. Προπαρασκευαστική δράση. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω διότι το αναφέρατε το θέμα αυτό και η σχετική ε, έκθεση έγινε. Όλα αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε αντικατοπτρίζονται στις, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Αυτή τη στιγμή συζητείται το χρονοδιάγραμμα με την ε, σχετική τροπή προϋπολογισμού. Όπως λέει ο δημοσιονομικός κανονισμός, το αργότερο, το τρίτον έτος της προπαρασκευαστικής δράσης, γιατί κάθε μία από αυτές διαρκεί περίπου τρία χρόνια, θα πρέπει η... το βασικό έγγραφο που αφορά ε, τους στόχους αυτής της δράσης να Υιοθετείτε και ελπίζουμε ότι στον επόμενη χρονική τρίτη περίοδο αυτό θα ισχύσει, αλλά δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει τίποτα συγκεκριμένο η επόμενο πρόγραμμα πριν από το, ε, να εκπνεύσει ορίζοντας 20.020. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή η προπαρασκευαστική ε, δράση θα ισχύσει στο 2018, 19 20. Και εδώ τίθενται, τίθενται διάφορα ε, προβλήματα. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αποδείξουμε κατά πόσο έχει προσθέμενη αξία η δράση αυτή. Άρα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε κάτι το επεφελές στα πλαίσια αυτής της ε, προπαρασκευαστικής δράσης, αλλά συζητούμε το θέμα, το όλο όπως σας είπα, διότι είναι θέμα κονδυλίων, με την ε, υπεύθυνη επιτροπή για θέματα, η διεύθυνση για θέματα προϋπολογισμού. Θα πρέπει λοιπόν ότι κάνουμε, το κάνουμε με μεγάλη προσοχή για να μην αποτύχουμε. Και αν δεν θέλουμε αποτυχία θα πρέπει να καταλήξουμε αφενός σε συμφωνία μαζί σας και από την άλλη με τα κράτη-μέλη και με την αμυντική βιομηχανία, πράγμα που δεν είναι το πιο εύκολο. Παρά το γεγονός ότι μετά από τις συζητήσεις που είχαμε μαζί τους, μπορώ να πω ότι ούτε μεταξύ τους οι διάφοροι φορείς της αμυντικής βιομηχανίας μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία. Αλλά σωστά αναφέρατε αυτά που είπατε. Αν θέλουμε όντως να δώσουμε πολιτική όθηση στην δράση που αναλαμβάνουμε σε πολιτικό ε, επίπεδο, θα πρέπει να κάνουμε κάτι που να φανεί ε, με σαφήνεια πριν από το 2016-2017. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντί. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δίστασα να ζητήσω το λόγο, μια που δεν είμαι τακτικό μέλος της Επιτροπής, έχοντας όμως συνεργαστεί με τον συνάδελφο Γκάλερ και τον ευχαριστώ για την τόσο σημαντική δουλειά που έχει κάνει προκειμένου να γνωμοδοτήσει στους ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων το Δεκέμβριο που έλαβε υπόψη του και την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, την οποία είχα αναλάβει εγώ. Όταν λοιπόν συζητήσαμε για αυτό το θέμα, όλοι οι συγητές από όλες τις πολιτικές ομάδες δεν ασχοληθήκαμε με το δημοσιονομικό ζήτημα, γιατί διαπιστώσαμε ότι κάθε φορά που μπαίναμε σε θέματα προϋπολογισμού, τότε φτάναμε σε διαφορετικές απόψεις που κινδύνευαν να θέσουν σε κίνδυνο την συνένεση προκειμένου να πάμε με συνένεση στην ε, Ολομέλεια. Έτσι λοιπόν τα θέματα τη δημοσιονομικά, το θέμα της χρηματοδότησης της επιστημονικής έρευνας για την αμυντική βιομηχανία ήταν πράγματα που αφήσαμε με την ιδέα ότι τα πράγματα στον τομέα αυτό προχωρούν πολύ όταν υπάρχει η ένοπλη σύραξη και πολύ λιγότερο όταν υπάρχει ειρήνη ενώ εμείς σκεφτήκαμε ότι και σε περίοδο ειρήνης πρέπει να προχωρούν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και συμφωνήσαμε μεταξύ μας να έχουμε πρώτα ε, συζήτηση στα πλαίσια των εκλογών του 2014, αλλά μετά Συμφωνήσαμε και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με το Συμβούλιο όταν αποφασίσαμε για το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 να υπάρξει πολιτική αναθεώρηση το 2016. Τη στιγμή δηλαδή που θα υπήρχαν νέα στοιχεία σημαντικά για τους ίδιους πόρους, ίσως και το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως τα κρατη κατά πάσα πιθανότητα να έχουν βάλει τάξη στα δημοσιονομικά τους, οπότε να είναι καλύτερα σε θέση να δεχτούν συνεισφορά για σχέδια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε λοιπόν την εντύπωση ότι η ιδέα αυτή θα μπορούσε να προχωρήσει. Δηλαδή να έχουμε προτάσεις ώστε ο προπολογισμό να είναι πιο σημαντικός για την επιστημονική έρευνα σε υλικά ή σε στρατιωτικές έρευνες ή μικτές και στρατιωτικές και μη στρατιωτικές και εν ώψη των εκλογών του 2014 αλλά και από το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο θα μπορούσε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσεις για να αυξηθεί ο προπολογισμό του ορίζοντα 2020 γιατί στην Ήτρε η δικιά μας έμονη ιδέα ήταν ότι δεν θέλουμε τα 70 δισεκατομμύρια του ορίζοντα 2020 να πειραστούν από επιπλέον δαπάνε. Αν όμω μπορούν να γίνουν πολιτικέ συζητήσει για να αυξηθεί ο συνολικό προπολογισμό, δεν πετύχαμε τα 100 δι που θέλαμε, αλλά ίσω τότε, αν έχουμε ε, μεγαλύτερα κονδύλια το 2006, να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια από την αύξηση αυτή και στο θέμα που συζητάμε. Πιστεύετε ότι έχει νόημα μια τέτοια πολιτική συζήτηση, θα ήταν χρήσιμη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριο Ντί. Παρακαλώ για να απαντήσετε. Χα, πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις αυτές που κάνετε τώρα λίγους μήνες πριν από το τέλος της θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θα απαντήσω στο τεχνικό σκέλος, γιατί η αναθεώρηση του 2016 του προπολογισμού είχε σαν σκοπό να απαντήσεις, στις κριτικές που έλεγαν ότι δεν είναι αρκετά ελαστικός ο προπολογισμό. Αυτή είναι η βασική ιδέα πίσω από την αναθεώρηση. Να δούμε μήπως πρέπει να γίνει ένα νέο χτένισμα ανάλογα με τις νέες προκλήσεις που θα έχει μπροστά της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει κατά τη γνώμη μου ότι μπορεί να υπάρξει αλλαγή χωρίς να αλλάζει η ίδια η φύση των χρηματοδοτικών μέσων το να βγει από ένα χρηματοδοτικό μέσο και να πάει σε ένα άλλο, ένα κονδύλι ή να μετακινηθούν χρήματα τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν σε κάποιο χρηματοδοτικό μέσο και να πάνε σε κάποια άλλα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία απορροφούν περισσότερα κονδύλια και όπου χρειάζεται πολιτική δράση, αυτό είναι πιθανό να γίνει. Υπάρχει δηλαδή περιθώριο ελιγμών για την αναθεώρηση το 2016. Αλλά είναι δύσκολο τώρα να πω αν το 2016 θα υπάρχει περιθώριο για πιο δραστική ή πιο μεγάλη αλλαγή στον προπολογισμό μας. Είναι νωρίς να το πω. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας λέει ότι τέτοιες θεμελιώδεις αλλαγές που απαιτούν ομοφωνία χρειάζονται χρόνο, διαπραγματεύσεις και είναι κάτι δύσκολο. Υπάρχει περιθώριο όμως να αυξηθεί ένα κονδύλι εφόσον μειωθεί κάποιο άλλο όπου η ζήτηση είναι χαμηλή, η απορρόφηση δεν είναι αρκετά μεγάλη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σοντή είναι ικανοποιημένο φαίνεται από την απάντησή σας. Έτσι. Δεν βλέπω να ζητάει κανένας άλλος το λόγο. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δουκάσκη. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, είναι και η τελευταία συνάντηση της Επιτροπή μας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε, τη σύμπτωση και ο τελευταίος προσκεκλημένος είναι Πολωνός και ο Προεδρεύων είναι Πολωνός. Λοιπόν, θα τελειώσουμε πολύ σύντομα και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Προέδρου μας, του κ. Ντανζό και του Προεδρείου της Επιτροπής αυτής, όλους σας για τη συμμετοχή σας την τελευταία πενταετία στην, στο έργο της Επιτροπής αυτής Ασφάλειας και Άμυνας. Ευχαριστώ πολύ επίσης όλους τους εκπροσώπους που έχουμε εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που πολύ συχνά ερχόσασταν στις συνεδριάσεις μας. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά, νομίζω, με όλους. Και με το ΝΑΤΟ και με την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Ευχαριστώ όλους τους προσκεκλημένους μας επίσης. Ευχαριστώ όλες τις πολιτικές ομάδες, τους συμβούλους τους, τους βοηθούς των Ευρωβουλευτών, όλους όσοι μας βοήθησαν να εργαστούμε καλά όλα αυτά τα χρόνια. Και όλος ιδιαιτέρως θέλω να ευχαριστήσω τη γραμματεία της Υποπιτροπής. Α, βέβαια, ξέχασα κάτι, ξέχασα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Εννοείται, η ΑΦΕΤ βασικά νομίζω θα έπρεπε να την ευχαριστήσει. Πάντως ευχαριστώ πολύ τη γραμματεία μας, όλα τα μέλη του προσωπικού της Υποπιτροπής αυτής δεν θα ήταν δυνατόν να δουλέψουμε τόσο καλά χωρίς τη δικιά σας παρουσία. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της Υποπιτροπής και όλων μας τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος, για την συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα πέντε χρόνια. And I have a pleasure. Και με πολύ χαρά. Α, ναι. Κάτι ακόμα για τους ευρωβουλευτές. Εύχομαι σε όλους σας, εφόσον είσαστε υποψήφοι, Καλή επιτυχία στις 25 Μαΐου. Και δεν μπορώ να σας δώσω την ημερομηνία της επόμενης συνεδριάσεώς μας, γιατί αυτό είναι κάτι που θα αποφασιστεί μετά τις ευρωεκλογές. Και πάλι σας ευχαριστώ. έλξη συνεδρίαση.